Η επόμενη Ολομέλεια θα διεξαχθεί αύριο στι 23 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 12. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγη συνεδρίασή μας. Καλό σα βράδυ.